Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής ως πρώτος αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μπορώ να σας καλωσορίσω σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτήν την τέταρτη κοινοβουλευτική εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα λέει και στα ελληνικά και στα γαλλικά ο πρόεδρος και στα ιταλικά. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ζαν Κλόντο Γιούνκερ, που ήρθε σήμερα εδώ. Ο κύριος Σούλτς, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι στο δρόμο. Έρχεται από το Λονδίνο. Θα είναι εδώ σε μισή ώρα. Είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κάμερον εκεί. Η Ολομέλεια αυτή λοιπόν κηρύσσει την έναρξη της 4ης Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας όπως είπαμε. Είναι μια διάσκεψη σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και αύριο θα λάβει χώρα συνάντηση για το άρθρο 13 όπου θα συμπροεδρεύει το Ολλανδικό Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών. Ο πρόεδρος Τούσκ θα είναι παρόν ε, από ό,τι φαίνεται σήμερα σκόπευε να είναι εδώ, αλλά ταξιδεύει ανά την Ευρώπη για να προετοιμάσει τις συζητήσεις που θα λάβουν χώρα στην διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτή τη βδομάδα. Συνεπώς, ο κύριος Τούσκο ζητά συγγνώμη για την απουσία του αυτή. Η συνάντηση αυτή πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντική για σας που είσαστε βουλευτές στα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά και για μας που είμαστε ευρωβουλευτές. Είμαστε φίλοι. Πρέπει να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, ποιοι είναι οι κανόνε για τη διεξαγωγή τη συνάντηση αυτή. Υπογραμμίζω ότι ω ήθιστε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ωστόσο γίνεται περισσότεροι συμμετέχοντε να μπορέσουν να εκφράσουν τι απόψει του εδώ. Ακόμα και αν έχουμε περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μα. Επειδή λοιπόν ακριβώ οι συμμετέχοντε είναι πάρα πολλοί, θα ήθελα να σα ζητήσω τι παρεμβάσει σα να τι περιορίσετε σε δύο λεπτά αναερώτηση στην ε, εξέλιξη τη συζήτηση. θα δούμε μήπω χρειαστεί να περιορίσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το χρόνο. Έχετε μπροστά σας κάτι κάρτες με τις οποίες μπορείτε να δηλώσετε ότι θέλετε να συμμετάσχετε στη συζήτηση, ότι θέλετε το λόγο. Οπότε όσο γίνεται πιο γρήγορα συμπληρώστε αυτές τις κάρτες και δώστε τις στους ε, κλητήρες. Και είναι σημαντικό να γίνει αυτό τώρα γρήγορα γιατί θα αλλάξω το πρόγραμμα και καλό θα ήταν να έχουμε 15-20 λεπτά με την παρουσία του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ερωτήσεις και απαντήσεις. Οπότε σας παρακαλώ, προετοιμαστείτε, συμπληρώστε την κάρτα αίτησης λόγου ώστε να μπορέσετε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα προσπαθήσουμε να χωρίσουμε το χρόνο ομιλία ως εξής. Δύο ή τρεις βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια, στη συνέχεια ένας Ευρωβουλευτής και ούτω καθεξής. Αν χρειαστεί θα προσαρμόσουμε όμως και αυτή τη φόρμουλα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 9 με 10 βουλευτές θα μπορέσουν να πάρουν το λόγο και μετά θα απαντήσει ο πρόεδρος Γιούνκερ και μετά θα μπούμε σε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων και θα απαντήσει ο κύριος Γιούνκερ και πάλι. Οπότε, θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο Γιούνκερ και μετά θα μπορέσετε να ρωτήσετε τον πρόεδρο Γιούνκερ. Και μετά θα ακούσουμε την ομιλία του κύριου Σούλτς. Παρακαλώ, κύριε πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει Πέμπτη και Παρασκευή. Γι' αυτό θα συναντηθώ σήμερα και αύριο με 21 πρωθυπουργούς. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι σε μισή ώρα θα πρέπει να καταλήψω την ε, συνάντηση αυτή και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, αλλά δεν ήταν δικιά μου ιδέα να οργανωθεί η συνάντηση αυτή αυτή τη βδομάδα, την ίδια με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και ελπίζω την επόμενη φορά που θα οργανωθεί αυτή η κοινοβουλευτική εβδομάδα να μην συμπέσει με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τόσο πολύ να κάνω ομιλία, αλλά θα ήθελα να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε, να ακούσω τις δικές σας παρατηρήσεις και τα δικά σας σχόλια. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο δεν είναι μια τεχνική διαδικασία, είναι κυρίως πολιτική και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπαγορεύει στις χώρες μέλη τι πρέπει να κάνουν, θέλει να ακούσει και γι' αυτό θέλω και εγώ να σας ακούσω αμέσως και μετά να μπορέσω να απαντήσω. Πρόεδρος Σταγιάννη. Ωραία. Περνώ στα γαλλικά τώρα. Και γιατί, γιατί η πρώτη ερώτηση είναι από την Γαλλική Εθνική Συνέλευση, κυρία Ντανιέλ Ρουά, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής για Ευρωπαϊκά Ζητήματα στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο ευθύ αμέσω. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, για να σα δω, δεν σας βλέπω, λέει ο πρόεδρο Γιούνκερ. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Λοιπόν, έλεγα ότι χαίρομαι που έχουμε αυτή την ε, κοινοβουλευτική εβδομάδα με διακοινοβουλευτική συζήτηση έτσι όπως αποφασίσαμε στο Λουξεμβούργο. Και είναι σημαντικό τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργάζονται όσο γίνεται περισσότερο στην αρχή της διαδικασίας αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Έχω δύο ερωτήσεις λοιπόν προς τον κύριο Γιούγκερ. Πρώτον, έχουμε την αίσθηση ότι δημιουργούμε την Ευρώπη του φόβου και η Ευρώπη της αλληλεγγύης και της πλήρους απασχόλησης δεν είναι τόσο ορατή. Ο τρόπος λοιπόν λειτουργίας που εφ' θα συμμετέχουν περισσότερο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι που είναι πιο κοντά στους πολίτες. Πιστεύετε ότι είναι ένα μήνυμα μπορεί να βοηθήσει. Και δεύτερον, για το ανανεωμένο ευρωπαϊκό εξάμεινο υπάρχει έλεγχος από τα κοινοβούλια και υπάρχουν τρεις κοινωνικοί δείκτες στα οικονομικά ζητήματα. Αυτή η προσθήκη βέβαια αμφισβητείται από κάποιους ε, βουλευτές. Εγώ είμαι υπέρ. Οπότε κύριε Πρόεδρε μπορείτε να μας διευκρινίσετε πώς εσείς βλέπετε αυτούς τους δείκτες και ποια είναι η άποψή σας για τους κοινωνικούς αυτούς δείκτες. Νομίζω ότι η δικιά σας άποψη θα δώσει περισσότερη, περισσότερο σώμα και περισσότερη ελπίδα σε αυτούς που υποφέρουν και ιδίω θα στηρίξει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Κύριε Γιούνκερ, να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, έχετε δίκιο. Η Ευρώπη του φόβου, η Ευρώπη του άγχους, της αγωνίας, όντως δημιουργείται αυτή τη στιγμή. Και ορισμένοι θέλουν να τροφοδοτούν τέτοιου είδους ε, αισθήματα. Που όμως είναι αρνητικά, είναι αρρωστημένα. Ανάμεσα στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της οποίας προεδρεύω, ξέρετε ότι έχουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση. Και κάθε άλλο παρά υπέρ μιας τυφλής λιτότητας είμαι. Και θα ήθελα να λυθούν ακόμα περισσότερο υπόψη διαστάσεις της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Γι' αυτό και από την αρχή της θητείας μας προτείναμε το ταμείο που πολλοί ονομάζουν Juncker, η ιδέα δεν ήταν να ονομάζεται έτσι, η ιδέα είναι να εντοπιστεί νομίζω, επειδή ονομάστηκε έτσι με το όνομά μου, να εντοπιστεί ο υπεύθυνο αν τυχόν αποτύχει. Αλλά δεν πρόκειται για αποτυχία. Διότι ήδη έχουμε κινητοποιήσει 61 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις 40 μεγάλα προγράμματα υποδομών έχουν αρχίσει ήδη σε 22 χώρες και δεκάδες χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επωφελούνται ήδη από αυτό το σχέδιο Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων με τη βοήθεια βέβαια και των κοινοβουλίων. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δίνω μεγάλη σημασία στην ε, συμβουλή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και ακριβώς γι' αυτό και χαιρόμαστε πολύ που είμαστε μαζί σήμερα το πρωί, γιατί το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη και συνενοχή θα έλεγα. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο στο βαθμό που μπορούν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια συνεργάζονται λοιπόν στενά όταν καθορίζονται οι μεγάλοι άξονες της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής. Επ' αυτού λοιπόν πρέπει επίσης να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα υπέρ των κοινωνικών δικτών. Εξάλλου το προτείναμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ΕΚΟΦΗΝ που απέριψε τους κοινωνικούς δείκτες που είχαμε εμείς προτείνει προς προβληματισμό στις εθνικές κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις λοιπόν σχεδόν με ομοφωνία απέρριψαν την ιδέα παρουσίας των κοινωνικών δικτών μεταξύ των εργαλείων μέτρησης της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλησης. Βέβαια δεν απελπίζομαι. Η κοινή λογική ελπίζω ότι θα περισχύσει. Και ότι και οι κυβερνήσεις θα ακολουθήσουν. Βέβαια, οι κυβερνήσεις πάνε πιο γρήγορα από την κοινή λογική μερικές φορές, αλλά νομίζω ότι θα παραδεχτούν κάποια στιγμή ότι χρειάζονται τέτοιοι δείκτε υπέρ τη δημοσιονομικής και οικονομικής σύγκληση και θα εξετάσουν όλα τα μέσα τα οποία μας επιτρέπουν να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα της κοινωνικής πραγματικότητας στην Ευρώπη, την οποία συχνά υποτιμήσαμε τις προηγούμενες χρονιές. Και γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει 8 Μαρτίου με μεγάλη διαβούλευση ακριβώς σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και τώρα από τη Λιθουανία η κυρία Μπιρούτε Μπερσάιτε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας ευχαριστώ πολύ για την ε, συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Όπως ε, γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή βιώνει πολλαπλές κρίσεις. Μετανάστευση, πρόσφυγες, παγκόσμια ανασφάλεια και έλλειψη εύρωσης οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. δεν ναι, γνωρίζετε ότι ο βασικός λόγος για την έλλειψη επενδύσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι η άνηση κατανομή του εισοδήματος. Τι πρέπει να κάνουμε. Δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στη δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά να αυξήσουμε και την αύξηση ε, σε εσωτερικό επίπεδο. Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ερώτησή μου βέβαια αφορά το εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που όταν γίνει το δημοψήφισμα το Μάιο ίσως ή δεν ξέρω πότε θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο αποφασιστεί το Brexit. Ε, πώς θα μοιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά ε, το Brexit αν όντω υλοποιηθεί. Ευχαριστώ. Κυρία μου, η παρέμβασή σας ήταν ε, δυτή. Το πρώτο τμήμα αφορούσε το επενδυτικό περιβάλλον στην Ευρώπη και το δεύτερο αφορά το ζήτημα της, του Ηνωμένου Βασιλείου. Για το πρώτο τμήμα της παρέμβασής σας θα ήθελα να πω ότι τα κράτη-μέλη που έχουν περιθώριο ελιγμών στον προπολογισμό τους θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν αυτά ώστε να μπορέσουν να δώσουν μια νέα ανάκαμψη στην ε, κατανάλωση. Διότι αν υπάρχει ιδιωτική κατανάλωση κατά τρόπον ώστε να μπορέσει ε, να συνδυαστεί με τις βασικές απαιτήσει στον προπολογισμό μπορεί να οδηγήσει σε ανάκαμψη. Αυτό που κάνουμε εμείς στα πλαίσια του, του σχεδίου επενδύσεων είναι τελείως διαφορετικό. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε ιδιωτικά κεφάλαια για να τροφοδοτήσουν τις δημόσιες επενδύσεις. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Το ερώτημα που θέτεται είναι διαφορετική φύσεως και έχει σχέση ε, με τις συγκεκριμένες συστάσεις αναχώρα που θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του Μαΐου την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε τις εκθέσεις αναχώρα και οι αξιολογήσεις που αναφέρεται θα περιλαμβάνονται στις διάφορες πρωτοβουλίες. Όσον αφορά τώρα το βρετανικό ζήτημα, θα συναντηθώ με τον Βρετανό Πρωθυπουργό εντός ολίγου. και μετά από τέσσερις με πέντε συναντήσεις ε, με τον ε, Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου διατύπωσε κάποιες προτάσεις, ε, διατυπώνουμε τις προτάσεις τις οποίες θα εξετάσουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή και θα δούμε εάν η απάντηση θα είναι καταφατική ή αρνητική. Θα δούμε δηλαδή αν οι προτάσεις του κυρίου Τούσκ και ε, του υποφαινόμενου θεωρούνται δίκαιες για τη Βρετανία και δίκαιες για, δίκαιες για τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη. Είναι πρόημο αυτή τη στιγμή να κρίνουμε το αποτέλεσμα. Αν σας έλεγα τώρα ότι έχουμε εφεδρικό σχέδιο, αυτό θα σήμαινε ότι υπάρχει διάθεση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ε, ε, προβλέψουμε ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει η Βρετανία από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε φεδρικό σχέδιο, έχουμε ένα σχέδιο Α. Η Βρετανία θα μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ενεργό και επικοδομητικό μέλος της. Και τώρα ο κύριος Πέδρος Σάουρα μέλος ε, του Κογκρές των Βουλευτών από την Ισπανία. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Η ερώτησή μου είναι για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά βάση, αλλά θα τη θέσω. Μεταξύ των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία σε οικονομικό επίπεδο κατά την άποψή μου είναι σημαντικά τα διαρθρωτικά προβλήματα, πάρα πολύ ε, σημαντικά, ε, η νέα μετριότητα, η κυκλική οικονομία και απαιτούν μεταξύ άλλων και ε, διεθνή συντονισμό στην οικονομία και στις οικονομικές πολιτικές. Υπ' αυτή την έννοια, κατά την άποψή μας, ο συντονισμός ε, σε θέματα φορολογίας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους τελευταίους αυτούς μήνες, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, προώθησε αρκετά πακέτα συντονισμού σε φορολογικά ζητήματα. Θα ήθελα λοιπόν να ε, ρωτήσω τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γιατί σας είπα ότι αυτό κυρίως αφορά αυτό τον ε, πρόεδρο του Συμβουλίου. Στην ε, τελευταία πρόταση του Επιτρόπου Μοσκοβισή είχαμε αυτές τις δύο οδηγίες, ε, συντονισμό σε διεθνές επίπεδο σε θέματα φορολόγησης, στρατηγική για τις ε, χώρες στις νέες συνθήκες που υπογράφονται για διπλή φορολόγηση δεν θα έπρεπε η το Συμβούλιο να μειώσει την φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτή τη ε, διεθνή συνεργασία. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί επιμένω ότι φρονώ ότι το οικονομικό πρόβλημα παγκοσμίω ε, δεν έχει να κάνει μόνο με συγκυριακά ζητήματα, αλλά και με διαρθρωτικά ζητήματα. Γι' αυτό υπάρχουν ε, φυσικά και μειώσεις και γι' αυτό χρειαζόμαστε και μια νέα πολιτική ε, αλλά χρειαζόμαστε πέραν της νέας πολιτικής και ε, διεθνή συντονισμό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βουλευτά, ο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών είναι μια πολύ ευρία έννοια και θα πρέπει φυσικά να βλέπουμε μακριά όταν συζητούμε το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών γιατί αποτελούν ε, τμήμα των οικονομικών πρακτικών και φυσικά έχουμε και τις ε, ε, δημοσιονομικές και φορολογικές πολιτικές γιατί για την Ευρώπη οποιαδήποτε τέτοια απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται ομόφωνα γι' αυτό και φυσικά υπάρχει πρόβλημα να προχωρήσουν αυτές οι υποτάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια πιο τολμηρή προσέγγιση σε θέματα συντονισμού ε, και για φορολογική εναρμόνιση. Έχουν γίνει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, κυρίως η, ένα σύστημα αυτόματων ανταλλαγών όσον αφορά τα tax rulings ε, και φυσικά και ένα σχέδιο δράσης ε, για τις διάφορες ε, πολιτικές σε θέματα φορολόγησης. Έχετε δίκιο βέβαια να πείτε ότι θα έπρεπε να είχατε αποφθεί το ερώτημά σας στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο πρέπει ε, να εξετάσει τις προτάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει να σας πω ότι εκ πρώτης όψεως οι προτάσεις μας δεν ε, ήταν προτάσεις οποίες αποδέχτηκαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό προτιμούν να ε, σταθούν σε δύο-τρεις χώρες αντί να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η Ευρώπη θα είχε κάνει πρόοδο αν είχε δεχτεί τις προτάσεις μας, κάτι το οποίο θεωρώ απαραίτητο. Έχουμε ακόμα πέντε ερωτήσεις. Ε, θα σας δώσω το λόγο και μετά θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο Γιούνκερ για να ολοκληρώσουμε. Ε, σας παρακαλώ λοιπόν να σέβεστε το χρόνο, ε, ένα λεπτό για την ερώτηση, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε και τη δυνατότητα στον πρόεδρο Γιούνκερ να απαντήσει. Η πρώτη ερώτηση είναι από τον κύριο Γιώακιμ Μπός από το Bundestag. Καλημέρα. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, σε αντίθεση με εσάς εγώ θεωρώ πως είναι ευτυχής η σύμπτωση αυτή την εβδομάδα ότι δηλαδή εμείς οι βουλευτές από τις χώρες της Ευρώπης μπορούμε τώρα να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για την κατάσταση στην Ευρώπη. Και αυτό μπορεί ίσως να οδηγήσει στο ότι θα ακουστούν και θα ληφθούν υπόψη σοβαρά αυτές οι ανησυχίες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ πως είναι ατυχής η συγκυρία γιατί είμαστε σε μια κατάσταση που δεν ε, έχει ξανασυμβεί τα τελευταία χρόνια και δεκαετίες. Τώρα, κάποιες ε, παρατηρήσεις. Πρώτον, υπάρχουν φήμες πως αρχηγοί σημαντικών ε, κρατών θέλουν να καθυστερήσουν την εμβάθυνση της Ένωσης. Αυτά τα οποία αναφέρατε δηλαδή στην έκθεση των πέντε Προέδρων μια περισσότερη σταθεροποίηση χωρίς αλλαγή των συνθήκων. Τι άποψη έχετε για αυτή την διαδικασία κύριε Γιονκέρ. Δεύτερον, ο πρόεδρος του S5, ο Ζίγμαρ Γκάμπριελ και οι υπουργοί οικονομικών χτες έγραψαν ένα άρθρο σε μια εφημερίδα στη Γερμανία και μίλησαν για την αναγκαιότητα η κάθε χώρα να κάνει αυτό το οποίο μπορεί ε, καλύτερα. Δηλαδή η Γερμανία να κάνει περισσότερες επενδύσεις. Αυτό όμως σημαίνει πως και άλλες χώρες θα πρέπει να δεχτούν πως χωρίς μια δικαιότερη κατανομή προσφύγων και μεταναστών δεν θα πετύχουμε την οικονομική σταθεροποίηση που θέλουμε. Υπάρχει μια σχέση μεταξύ αυτών των πραγμάτων που δεν την βλέπουν όλα τα κράτη. Και τρίτον για το φορολογικό ντάμπινγκ. υπάρχει Ολλανδική Προεδρία και είναι μια καλή ευκαιρία για τους Ολλανδούς να επιτύχουν κάποια πρόοδο, να αλλάξουν το οικονομικό τους μοντέλο και να συνεισφέρουν ε, στην μάχη κατά του φορολογικού ντάμπινγκ στην Ευρώπη. Τον λόγο τώρα... Έχει η κυρία Ερένα Γαρίδο από την Ισπανική Βουλή, από το Κογκρέσο των Βουλευτών. Ε, καλημέρα σας. Καταρχάς, ε, πολύ σύντομα να σας ευχαριστήσω που με επιτρέπετε να συμμετέχω ενεργά σε αυτή τη συνεδρίαση ε, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και η ερώτησή μου απευθύνεται στον κύριο Γιούνκερ. Εδώ και λίγες μέρες Έγινε μια σύντομη ε, σύνοψη των όσων πέτυχε το Στρατηγικό Ταμείο Επενδύσεων. Ε, είχαμε 200 ε, εκατομμύρια σε υποδομές, 84 σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Η Ισπανία έχει έξι προγράμματα. Και θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Με ποιο τρόπο η επιβράδυνση της ανάπτυξης θα επηρεάσει την εκτέλεση ε, και μάλιστα την ταχύτερη εκτέλεση αυτού του προγράμματος. Σας ευχαριστώ πολύ. now, Ο κύριος Γεράσιμος Μπαλαούρας τώρα, μέλος της Ελληνικής Βουλής. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, ε, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση, δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η Ευρώπη με μόνο μελιτότα, με δείκτες μόνο οικονομικούς, αγνοώντας τους κοινωνικούς δείκτες. Και μάλιστα όταν τα φάρμακα που επιπλέον προτείνουν είναι αυτά που σαπίζουν κομμάτια του οργανισμού. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εννοώ τους 1,5 εκατομμύρια ανέργους στην Ελλάδα, τα 3,5 εκατομμύρια στα, στα όρια της φτώχειας και τους χιλιάδες άνεργους στους δρόμους να κοιμώνται με κρύο και με βροχή. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Την υπενυχτήκατε κύριε Πρόεδρε. Ότι όταν τσακώνονται τα βουβάλια, λέμε στη χώρα μου, τα πληρώνουν τα βατράχια. Και ότι υπάρχει με διαφωνίες είτε μεταξύ των τριών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με, την, ε, με το Δούνου του, είτε και μεταξύ τους. Επίσης τώρα πάνω σε αυτή την αρρωστημένη κατάσταση προσ, ε, προσθέθηκε το προσφυγικό που στην Ευρώπη του διαφωτισμού, στην Ευρώπη της ανεκτικότητας και δημιουργούνται ξενοφοβικές καταστάσεις έντονες και θέλουν να, αρθώσουν, να ορθώσουν σύνορα, σύνορα που πώς μπορεί να σταματήσουν τις χιλιάδες τα εκατομμύρια ανθρώπους που θέλουν να φύγουν από ένα πόλεμο που και εμείς και κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευθύνονται. Υπάρχει λοιπόν πρέπει να γίνει μια βαθιά στροφή. Μια βαθιά στροφή στην κοινωνία με συλλογικότητα, με κοινωνικότητα και με ανθρώπινο πρόσωπο. Θέλω να πω τελευταίο ότι το Ευρωκοινοβούλιο, ακούγοντας και τους συναδέρφους που, που τους προλαλήθαντες, θεωρώ ότι πρέπει να αναβαθμιστεί. Να αναβαθμιστεί και όχι να είναι τύπης δημοκρατία, όχι μόνο να έχουμε μία φορά το εξάμεινο ή και οι ευρωβουλευτές ακόμα να έχουν ελάχιστε δυνατότητες παρέμβασης και να μεταφέρουν τις απόψεις, τα αισθήματα και τις αγωνίες των κατοίκων των χωρών που εκπροσωπούν. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. And now from... Σας ευχαριστώ από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ε, Βουλή των ε, Λόρδων η Βαρόνη Φόκνερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που δέχεστε και ερωτήσεις. Έχω κάποιες σύντομε ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ που δεν έχετε εναλλακτικό σχέδιο για το Brexit. Ελπίζω. Εμείς από τη δικιά μας ε, τη Σκοπιά ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Η Επιτροπή μας ε, συντάσσει μια έκθεση για την έκθεση των πέντε πρόεδρων και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Θεωρείτε πως ε, είναι εφικτά αυτά τα οποία λέτε στην έκθεσή σας γιατί είμαστε 8 χρόνια ήδη σε ύφεση και έχετε ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2025. Επίσης μιλάτε για διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Και με χαρά μιλάω μετά τον Γερμανό συνάδελφο γιατί η χώρα τους ε, βεβαίως είναι μια από τις χώρες που έχει υπερβολικό πλεόνασμα. Θεωρείτε λοιπόν πως έχετε κάποιες, ε, κάποια μέσα για να αντιμετωπίσετε τα υπερβολικά πλεονάσματα πέρα από τα ελλείμματα. Και τέλος, προβλέπετε κάποιο Υπουργείο Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ε, τελικό αποτέλεσμα της ε, Δημοσιονομικής Ένωσης με βάση τα όσα είπατε για τη σύγκληση. Σας ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση προς τον Πρόεδρο της Κομισιόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία Ροντρίγκε έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που ήρθατε. Όντως είναι δύσκολη η συγκυρία για όλου μα και για εσά. Εγώ μιλώ ω εισηγήτρια εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκθεση όσον αφορά την ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη. Συζητούμε ακόμα, όμω εγώ πιστεύω, έχω την πεποίθηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει μια έκθεση όπου η οικονομική και η κοινωνική σύγκληση προς τα πάνω θα είναι ο κεντρικός στόχος όπως το πρότεινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξάλλου. Αυτό σημαίνει ότι θα συμφωνήσουμε για το ότι οικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Και αυτό σημαίνει με τη σειρά του ότι για να το στηρίξουμε πρέπει να προχωρήσουμε με το σχέδιο επενδύσεων και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις υπέρ των επενδύσεων και της απασχόλησης. Εμείς πιστεύουμε ότι η ανάκαμψη, η οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη έχει κεντρικό ρόλο για να επιτευχθεί η συνοχή στην Ευρώπη μεταξύ των Ευρωπαίων και να βοηθήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές ε, κρίσεις που βιώνει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν πιστεύω ότι πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Είμαι πεπισμένη ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά με τα Εθνικά Κοινοβούλια και από εκεί και πέρα αυτό που θέλω να μάθω είναι κατά πόσο μπορούμε από κοινού να αρχίσουμε να εργαζόμαστε πιο συστηματικά πια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε το πλοίο να πάει προς την ίδια κατεύθυνση. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Δίνω το λόγο στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλόντο Γιούνκερ, για να απαντήσει στις ε, ερωτήσεις σας και να ολοκληρώσουμε αυτό το τμήμα που έχει να κάνει με τις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια και την Κομισιόν. Γιούνκερ. Πρόεδρε, υπάρχουν συνάδελφοι λοιπόν πέντε που έθεσαν ερωτήσεις, αλλά έθεσαν 14 ερωτήσεις συνολικά. Λοιπόν, ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας ε, είναι λίγος, γι' αυτό θα απαντήσω στους πέντε συναδέρφους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον συνάδελφο πώ. ο οποίος διαπίστωσε πως υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί και κάποιοι λιγότερο σημαντικοί ηγέτες ε, κρατών. Δεν ξέρω ποιους εννοείται σημαντικούς, ε, γιατί δεν ξέρω, εγώ τους θεωρώ όλους σημαντικούς ή ασήμαντους βεβαίως, αναλόγως. Λοιπόν, θεωρώ πως η έκθεση των πέντε πρόεδρων είναι μια πρόταση των ε, πρόεδρων θεσμικών οργάνων που πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά ε. γιατί θεωρώ πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να έχουν λόγο γι' αυτό ακριβώς συμμετείχε ο πρόεδρος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την έκθεση γιατί βεβαίως ε, δεν θα είχε και αυτή τη μορφή η πρότασή μας. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρές ε, διαφορές απόψεων μεταξύ σημαντικών και μη, όπως είπατε, αρχηγών κρατών όσον αφορά την εγγύηση των καταθέσεων, αλλά υπάρχουν κάποιοι αρχηγοί κρατών οι οποίοι δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν αμέσως, κυρίως ε, γιατί θεωρούν πως ε, υπάρχει κάποια ιστεροβουλία στην πρότασή μας ε, αυτή. Δεν είναι ότι λέμε ότι ξαφνικά θα υπάρχει μια πανευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων από τη μια μέρα στην άλλη. Όχι, υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν. Δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά από το 2024 και όπως είπα ε, θα πρέπει να γεμίσουν τα ανάλογα εθνικά ταμεία να το πω έτσι πριν μπορέσει κανείς να ζητήσει την ευρωπαϊκή βοήθεια σε αυτό το θέμα. Επίσης με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο περισσότερων εθνικών ε, και περιφερειακών ε, επενδύσεων. Βεβαίως αυτό δεν είναι αποστολή της Κομισιόν, αλλά θα καταθέσουμε κάποιες σχετικές ε, προτάσεις προσεχώς για να κλείσει αυτό το κενό των επενδύσεων. Ειδικά στον, στο επίπεδο των δήμων και των περιφερειών. Ξεκολουθούμε Ξέρετε πως ε, αυτή τη στιγμή οι Δήμοι ε, κατά μέσο όρο 70% λιγότερο από ό,τι έκαναν το 2008. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποια αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος ε, και υπάρχουν βεβαίως και σχέσεις ε, με την εκτέλεση του υπολογισμού, όπως είπατε με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και με το θέμα των ε, προσφύγων ε, και μεταναστών. Πράγματι πρέπει να το δούμε αυτό. Τώρα το θέμα το οποίο είπατε για την για το φορολογικό dumping. Αν θυμάμαι καλά, η Κομισιόν έχει κάνει τις ε, προτάσεις που έπρεπε και πράγματι η Ολλανδική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή εργάζεται προς την εφαρμογή τους ε, και η Ολλανδική Προεδρία νομίζω πηγαίνει προς έναν ε, συντονισμό αν όχι μια εναρμόνιση των φόρων στην Ευρώπη. Μια άλλη ερώτηση από μια συνάδελφο Ισπανίδα νομίζω, είχε να κάνει με το πόσο γρήγορα θα τεθεί σε εφαρμογή το επενδυτικό σχέδιο. Είναι αλήθεια ότι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μπορέσαμε να κινητοποιήσουμε έναν, ένα μεγάλο ποσό ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων με αποτέλεσμα έργα σε 22 χώρες υπέρ πολλών μικρών και μεσαίων επενδύσεων. Βέβαια, η ανάπτυξη παραμένει χαμηλή, αλλά δεν θα το συνδέσω άμεσα με το σχέδιο. Θα έλεγα ότι όσο πιο αδύναμη είναι η οικονομική ανάπτυξη, τόσο πιο μεγάλη πρέπει να είναι και η πρόθεσή μας να εφαρμοστεί γρήγορα το επενδυτικό σχέδιο και που δεν θα πρέπει να περιοριστεί στα τρία επόμενα χρόνια, θα πρέπει να παραταθεί θα έλεγα εγώ, και στην επόμενη περίοδο θητείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για, τους, για τον Έλληνα συνάδελφο θέλω να πω ότι εγώ δεν είμαι υπέρ και το έχω πει και το έχω αποδείξει της λιτότητας, της τυφλής λιτότητας. Διαφωνώ με την ιδέα ότι η απάντηση στην κρίση είναι η λιτότητα, η υπερβολική λιτότητα. Όχι. Εγώ είμαι υπέρ του μείγματο της βελτίωσης των δημοσιονομικών μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εξετάζονται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ακριβώς και επενδύσεων. Χρειάζονται όλα αυτά τα στοιχεία για να έχουμε ένα καλό μείγμα στις ευρωπαϊκές μας πολιτικές. Και δεν είμαι και υπέρ του κλεισίματος των συνόρων. Εγώ βρίσκω ότι είναι ανόητο. Επειδή δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος των εξωτερικών μας συνόρων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει προτάσεις να παρετούμαστε. Μα ή που είμαστε μία ήπειρος ή που είμαστε ένα σύνολο το οποίο διαιρείται σε εθνικές κατηγορίες. Κάτι πολύ αρνητικό και που δυστυχώς το κάνουν κάποιες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις ήδη από τον Ιούλιο του 2014. Προτείναμε την επανεκατάσταση των ε, προσφύγων που ήδη βρίσκονται στην επικράτειά μας. Να τους μεταφέρουμε δηλαδή και να τους μοιράσουμε στις διάφορες χώρες. Προτείναμε για τα εξωτερικά σύνορα και προτείναμε κοινό διάβημα από όλε τις χώρες ε, μέλη όσον αφορά τις ε, χώρες προέλευσης. Αν είχαν γίνει όλα αυτά που είχαμε προτείνει, η κατάσταση σήμερα θα ήταν πολύ καλύτερη από αυτή την χαοτική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Κύριε Ροντρίγκε, συμφωνώ μαζί σας και έτσι έχουν τα πράγματα εδώ και έναν αιώνα. Δυστυχώς πρέπει να φύγω τώρα, να αποχωρήσω. Σας αφήνω στα αδέξια χέρια του Προέδρου λέει ο κ. Γιούνκερ χαριτολογώντας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Οι απαντήσεις σας ήταν πολύ ενδιαφέρουσε για όλους εμάς και ιδιαίτερα αυτά τα τελευταία που είπατε για τη σχέση του πρώτου πυλώνα, δηλαδή επίλυση του θέματος του χρέους, με το δεύτερο πυλώνα που είναι ανάπτυξη. Ευχαριστούμε πολύ Πρόεδρε για το διάλογο αυτό. Καλή τύχη στη συνέχεια και καρποφόρες εργασίες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Σούλτς, έρχεται και πριν από την ε, ομιλία του και την ολοκλήρωση του πρώτου τμήματος της συνεδριασής μας, θα ήθελα να σας ενημερώσω λίγο για το σημερινό πρόγραμμα. Μετά την ε, πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας θα γίνει μια δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας η οποία θα είναι αφιερωμένη στις ε, πολιτικές προτεραιότητες ε, του κύκλου αυτού του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα γίνει εδώ σε αυτή την αίθουσα. θα προεδρεύει ο κύριος Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη, πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο Τόμας Χάντελ, πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτή τη δεύτερη συνεδρίαση θα είναι παρόν και ο ε, Βάλτης Ντομπρόσκης, αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρώ και το Κοινωνικό Διάλογο και ο Πιέρ Μοσκοβισή, Ευρωπαϊο Επίτροπο για τα οικονομικά και νομισματικά θέματα, τη φορολογία και τα τελωνία. Θα γίνει διάλειμμα στη συνέχεια μεταξύ 1 και 3 και θα παρατεθεί γεύμα. Ε, από τη 1 ω τι 3 θα συνεδριάσουν οι πολιτικέ ομάδε και στι 3 η ώρα το απόγευμα θα συνεδριάσουν οι διακοινοβουλευτικέ επιτροπέ και εδώ έχουμε συνεδριάσει στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Θέμα θα είναι η παρακολούθηση ε, ε, των ΠΕΠΣ ε, στην αίθουσα PHS 3C050. Είναι ακριβώς απέναντι από την Ολομέλεια. Η δεύτερη συνεδρίαση που οργανώνεται από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ε, με θέμα ε, τι είναι ένα κοινωνικό ε, τριπλό α και έχουμε μηχανισμούς για την, ο καθορισμό των κοινωνικών δημοκραμάτων και των μισθών καθώς επίσης και μια τρίτη συνεδρίαση, ε, συγγνώμη, η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα Γιάν 4Q1 στο κτίριο Ζωζε Φαντάλ στο τέταρτο όροφο. Και επίσης έχουμε και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Το θέμα είναι ε, προσδοκίες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και τι ακριβώς θα γίνει με τις επόμενες διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο στην αίθουσα Γιάν 6Q2, κτίριο Ζωζε Φαντάλ, στον εκτό όροφο. Να σας επαναλάβω επίσης ε, στα γαλλικά, αυτά τα οποία είπα και στα, ελληνικά, ε, στα αγγλικά στην αρχή, όποιος επιθυμεί να θέσει ερωτήσεις θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο αυτό και να το παραδώσει στους κλητήρες. Α, πρέπει να γράψετε αν είστε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Εθνικού σας Κοινοβουλίου, το όνομα τεπώνυμό σας και ε, ε, το πολιτικό σας ε, κόμμα. Αν έχετε ρωτήσεις είτε για τον πρόεδρο Σούλτς είτε στη συνέχεια για τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Ντομπρόσκης ή τον επίτροπο, τον κύριο Πιέρ Μουσκοβισή. Θα έλεγα ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία. Ορισμένες φορές ε, είχα την εντύπωση ότι υπάρχει μία ε, διαμάχη μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Α, δεν είναι όμως αυτός ο κατάλληλος τρόπος να ερμηνεύουμε τις συνθήκες. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε διότι η νομοθετική δραστηριότητα και η επικουρικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Η νομοθετική δραστηριότητα ε, ξέρετε ότι όταν υπάρχει κάτι το οποίο αντιβαίνει στην επικουρικότητα και στις σχέσεις μεταξύ ημών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ημών από τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι πάρα πολύ σημαντικά και ιδίω όταν βιώνουμε χαλεπούς καιρούς για την ευρωπαϊκή οικονομία. Βιώνουμε κρίση, υπάρχουν πολύ επικίνδυνες προκλήσεις, η τρομοκρατία, επομένως θα πρέπει να λύσουμε και τα προβλήματα αυτά, τα θέματα της μετανάστευσης. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε όλοι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις στου συμπολίτε μας. Ε, και όσον αφορά την επικουρικότητα, ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς σεβόμαστε απόλυτα όλα τα εθνικά κοινοβούλια, ε, κοινοβούλια. Η έννοια τη επικουρικότητα είναι πολύ σημαντική. Ό,τι μπορέσετε να κάνετε εσείς ε, στο πλευρό των πολιτών είναι πολύ σημαντικό όπως είναι και για εσά φυσικά. Ε, θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία και όπως σας έλεγα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις στις διάφορες χώρες μέλη. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει. Η οικονομική κρίση ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Εχθές ε, συναντήσαμε εδώ τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Ντράγκη, ο οποίος είπε ότι πρέπει να συνεχίσουμε και η κατάσταση θα προχωρήσει πολύ αργά Πρέπει λοιπόν να γίνουν επενδύσεις και πρέπει να μπορέσουμε να μειώσουμε και τις δημοσιονομικές πιέσεις. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και για τους νέους μας, για το μέλλον. Υπάρχουν αρκετές προκλήσεις και θεωρώ ότι η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, που είναι και το μόνο ερετό όργανο μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και των Εθνικών Κοινοβουλίων πρέπει να ενισχυθεί γιατί εγώ θεωρώ ότι όλες μας οι συνεδριάσεις είναι πολύ σημαντικές. Επίσης, πρέπει να γίνονται συνεδριάσεις στις οποίες ε, θα υπάρχει μια διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήρθε και ο Πρόεδρος, του δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο για να ολοκληρώσουμε την πρώτη συνεδρίαση. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν ο Πρόεδρος ε, θέλει να απαντήσει στις ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Ταγιάννη. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, για την υπομονή σας και την παρουσία σας. Ζητάω συγγνώμη για την καθυστέρηση να ευχαριστήσω τον Αντώνιο Ταγιάννη για το ότι τελευταία στιγμή με αντικατέστησε. Και θα σας εξηγήσω γιατί δεν ήμουν εδώ στην αρχή αυτής της ε, συνεδρίασης. Ε, 9 με 10 είχαμε εδώ τον Βρετανό Πρωθυπουργό για να προετοιμάσουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον αναμέναμε αλλά λόγω τεχνικών δυσκολιών δεν ήταν εδώ πέρα στις 9 ήρθε στις 9.30 και ξεκινήσαμε τις συζητήσεις ε, λίγο πιο μετά, κράτησαν και λίγο παραπάνω. Οπότε ζητώ την κατανόησή σας για το ότι δεν ήμουν εδώ στην έναρξη. Έπρεπε να συζητήσουμε με τον κύριο Κάμερον για την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Πέμπτη στις ε, διαβουλεύσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το εάν θα παραμείνει η Μεγάλη Βρετανία στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, ε, ήρθα βεβαίως γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η συζήτηση και επαφή των Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι βεβαίως στο πλαίσιο του άρθρου 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, ούτως ή άλλως και αφορούν και τα ζητήματα τα οποία συζήτησα σήμερα το πρωί με τον Πρωθυπουργό τον κύριο Κάμερον. Γι' αυτό νομίζω πως ε, θα σας ενδιαφέρει και εσάς ε, να σας πω νολίγιστο ότι συζητήσαμε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Ξέρετε πως η Βρετανική κυβέρνηση θα ήθελε στην συνθήκη ε, να αλλάξει η διατύπωση η οποία μιλάει για μία ολοένα πιο στενή ένωση λαών. Αυτό αναφέρεται ως ε, στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κάτι το οποίο βεβαίως θεωρούν οι Βρετανοί ότι δεν τους δεσμεύει και θέλουν να αλλάξει η διατύπωση στην επόμενη αναθεώρηση της συνθήκης. Αυτό συζητήσαμε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό και οπωσδήποτε θα μας απασχολήσει και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γιατί υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη, νομίζω η πλειοψηφία ε, όπως και η πλειοψηφία νομίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν διαφορετική άποψη θεωρούν πως ε, κάποιους ε, τομείς πολιτικής που θα συζητήσετε και εσείς τις επόμενες ώρες χρειαζόμαστε στενότερη συνεργασία αν δούμε τις εξελίξεις στον τομέα των χρηματαγορών στον τομέα των τραπεζών νομίζω πως χρειαζόμαστε μια όλο ένα στενότερη ένωση και όχι να υπάρχει μια όλο και περισσότερη απομάκρυνση των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι δύο διαφορετικές θέσεις λοιπόν οπωσδήποτε θα συζητηθούν την πέμπτη που μας έρχεται και υπάρχει μια σειρά κρατών μελών και η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θεωρούν πως ε, δεν μπορεί σε μια μελλοντική αναθεώρηση της ε, συνθήκης ε, να είναι η μοναδική αλλαγή αυτή η φράση του Ever Closer Union. Θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Και βεβαίως αυτό θα πρέπει να περιέχεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το άλλο θέμα το οποίο συζητήσαμε ήταν οι σχέσεις της Ευρωζώνης ε, με τις ε, χώρες ε, μέλη που δεν είναι στο ευρώ. Είναι λοιπόν στην κοινή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζεται στις συνθήκες και είναι απολύτως θεμητή η τοποθέτηση νομίζω του Ηνωμένου Βασιλείου να μην υφίσταται κάποια διακριτική, δυσμενή μεταχείριση επειδή δεν είναι μέλος της Ευρωζώνης, ε, να μην υφίσταται δυσμενή μεταχείριση στο πλαίσιο της ε, κοινή αγοράς. Εξάλλου πρόκειται για μια χώρα που είναι καθαρός εισφορέας, συνεισφέρει πάρα πολύ στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, είναι σημαντικό κομμάτι της εσωτερικής αγοράς και θεωρώ πως ε, είναι απολύτως θεμητό να λένε πως δεν θέλουμε να έχουμε κάποιο μειονέκτημα στην εσωτερική αγορά μόνο και μόνο επειδή λάβαμε την απόφαση να μην μπούμε στο ευρώ. Νομίζω πως αυτό είναι απολύτως ε, θεμητό. Αλλά απ' την άλλη είναι και θεμητό τα κράτη της Ευρωζώνης να πούν πως μια εμβάθυνση της ε, Ευρωζώνης και οι αποφάσεις που λαμβάνουμε στην Ευρωζώνη δεν είναι δυνατόν να περιμένουν την έγκριση κρατών ε, εκτός της Ευρωζώνης. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν η μία πλευρά λέει δεν θέλουμε να έχουμε δυσμενή μεταχείριση αλλά να έχουμε βέτο στις αποφάσεις που λαμβάνετε εσείς. Και ακριβώς αυτό συζητήσαμε. Είμαι αισιόδοξο ότι την Πέμπτη θα υπάρξει σε αυτό κάποιος ε, συμβιβασμός. Επίσης, είναι ξεκαθάρισα πως ε, βάση και της εσωτερικής αγοράς και της ε, Ευρωζώνης είναι η συνθήκη. Στο άρθρο 3, παράγραφος 4, ξεκαθαρίζουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, έχει συστήσει μια ΟΝΕ, το νόμισμα της οποίας είναι το ευρώ και βεβαίως έχει το opt-out η Βρετανία και η Δανία. για τα λοιπά όμως κατά λοιπά ισχύει η συνθήκη και η συνθήκη προβλέπει πως οι χώρες οι οποίες δεν είναι στο ευρώ και δεν έχουν αυτή την ειδική πρόβλεψη όπως η Δανία και η Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει κάποια στιγμή να ε, υιοθετήσουν το κοινό νόμισμα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε την κατάσταση την εξή. 19 χώρες τη Ευρωζώνης, 7 τις οποίες αφορά η συνθήκη και 2 οι οποίες έχουν εξαιρεθεί. Και αυτό νομίζω θα αποτελέσει αντικείμενο συμφωνία την Πέμπτη και τέλος. Συζητήσαμε το θέμα της καλύτερης ε, συνεργασίας των θεσμικών οργάνων με τα εγώ υπενθύμησα πως ε, εδώ και ένα χρόνο περίπου τα τρία θεσμικά όργανα, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Κομισιόν διαπραγματεύονται μια διοργανική συμφωνία μεταξύ τους για την καλύτερη νομοθεσία όπως ε, λέγεται και υπάρχει εδώ πέρα μια μεγάλη λίστα απαιτήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για τη μείωση των επιβαρύσεων στις μικρές και μισές επιχειρήσεις, για την κατάργηση περιτών ρυθμίσεων, για την μείωση του διοικητικού άχθους των διατάξεων αυτών και διαφόρων κανόνων που πραγματικά ε, κάπου τους ε, ενοχλούν και σε αυτά συμφώνησε ούτως ή άλλως και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία και νομίζω πως ε, έχουν γίνει δεκτά σε μεγάλο βαθμό πριν πάμε καν στο Συμβουλίο και υπάρχει και το τελευταίο θέμα το οποίο οπωσδήποτε μας απασχολεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια το ζήτημα των λεγόμενων κοινωνικών ε, επιδομάτων στα κράτη-μέλη πώς μπορούμε να αποφύγουμε την κατάχρησή τους αφενός αλλά ταυτόχρονα να μην εμποδίσουμε την ελεύθερη κινητικότητα των πολιτών, των εργαζομένων στην εσωτερική αγορά και να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο γιατί υπάρχουν δύο αρχές οι οποίες ε, συγκροτούνται και οι οποίες βεβαίως δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Υπάρχει στην εσωτερική αγορά εγγύηση της ελεύθερης μετακίνησης, κάτι το οποίο σημαίνει πως οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εγκατασταθούν, να εργαστούν σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης. Και κανένας ε, δεν θα πρέπει να υφίσταται κάποια διάκριση λόγω της ε, υπηκότητας, ε, θρησκείας, χρώματος κτλ και βεβαίως οπωσδήποτε λόγω της ε, χώρας προέλευσης. Από την άλλη βεβαίως είναι λογικό ε, ένα κράτος να αισθάνεται πως ε, όταν ε, υπάρχει συστηματική εκμετάλλευση του κράτους προνοίας που έχει δημιουργήσει να μπορεί να αμυνθεί απέναντι σε αυτό χωρίς βεβαίως να υπάρχει διακριτική μεταχείριση Ευρωπαίων πολιτών. Τα συμπεράσματα λοιπόν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αφορούν την νομοθεσία. Στην ε, νομοθεσία αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης μαζί με το Συμβούλιο και υπενθύμησα πως θα επιμείνουμε στην τήρηση των αρχών που αναφέρονται στην συνθήκη. Αυτό σας αφορά οπωσδήποτε και στις χώρες σας γιατί ε, Οπωσδήποτε επηρεάζονται τα κοινωνικά συστήματα και στις χώρες σας από αυτή την συζήτηση. Αυτά λοιπόν ήταν τα βασικά σημεία τα οποία συζητήσαμε και τα ανέφερα γιατί ως γνωστόν είμαστε διατεθειμένοι να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να μην διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να παραμείνει μέλος η Μεγάλη Βρετανία. Εγώ τουλάχιστον παλεύω γι' αυτό και θεωρώ πως είμαστε χειρότεροι με τη Μεγάλη Βρετανία αλλά και η Μεγάλη Βρετανία είναι ισχυρότερη ως ε, μέλος της Ένωσης και ως γνωστόν ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και είναι κάτι το διαφορετικό το να υπάρχει μια γενική εκδήλωση της ε, βούλησής μας με το πώς μεταφράζεται αυτό στην πραγματικότητα και στις ε, λεπτομέρειες. Νομίζουμε λοιπόν, ξέρετε ότι θα διεξαχθεί και ένα δημοψήφισμα και υπάρχει βεβαίως και το ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει την πέμπτη των προσφύγων αλλά και το θέμα της Συρίας και των τελευταίων εξελίξεων που είναι ανησυχητικές ε, αυξάνονται οι συγκρούσεις ε, αυξάνονται α, τα θύματα μεταξύ των αμάχων και θα πρέπει όλοι να φροντίσουμε να μην υπάρξει περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Αντιθέτως όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να διαπραγματευτούν στη Γενέβη χωρίς ε, προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν θα υπάρξει στρατιωτική λύση στην Σύρια. Γιατί βλέπω πως ε, θα είναι εδώ πέρα και η τουρκική κυβέρνηση παρούσα την Πέμπτη και θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε μαζί τους ε, και το θέμα των προσφύγων αλλά και το θέμα της αποκλιμάκωσης της στρατιωτικής δράσης ε, στη Συρία. Ανέφερα αυτά τα πράγματα εν Ξέρω πως δεν είναι στην ημερήσια σας ε, διάταξη αλλά δεδομένης της κατάστασης και της καθυστέρησής μου νομίζω πως ε, λογικό ήταν να μάθετε γιατί καθυστέρησα και ο κύριος Γιούνκερ νομίζω σας εξήγησε ήδη πόσο ε, σημαντική θεωρούμε την ε, συνεδρίαση αυτή ο κ. Σταγιάννη δεν ήξερε ότι θα προεδρεύσει το πρωί που τον ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και Ευχαριστώ και σας για την προσοχή σας. There are eight... Έχω 8 μιλητέ στον κατάλογο. Ένα λεπτό ο καθένας παρακαλώ. Και στη συνέχεια ο πρόεδρος Σούλς θα απαντήσει για να ολοκληρώσουμε την συζήτηση αυτή. Ο πρώτος από την Αυστρία. Ο κύριος Κράινερ. Παρακαλώ. Uh, yes, thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να επανέλθω στη συζήτηση που είχαμε πριν. Οι χώρες που έχουν όντως πλεόνασμα στον προπολογισμό τους πρέπει να το χρησιμοποιήσουν, μπορούν και πρέπει για να ενισχύσουν τη ζήτηση. Δεν νομίζω όμω ότι το θέμα της ιδιωτικής κατανάλωσης είναι το πρόβλημα στην Ευρώπη μόνο, είναι οι επενδύσεις, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικέ. Αν λοιπόν λέμε τι μέγεθος πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα που να μπορεί να βασιστεί στα πλεονάσματα, θα πρέπει να είναι ένα ευρωπαϊκό 1% του ΕΠ θα έλεγα τότε μιλάμε για 130-140 δισεκατομμύρια. Ενώ τώρα είμαστε στα 4-6. Όχι ότι δεν θεωρώ ότι είναι θετικό το σχέδιο Juncker, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο και ήρθε πολύ αργά. Και να πω δύο λόγια και για την προσφυγική κρίση, παρακαλώ. Δεν είναι μόνο τρεις χώρες στην Ευρώπη που μπορεί να θεωρηθούν είναι οι υπεύθυνε που έχουν βοηθήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που φεύγουν από τον πόλεμο, είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Και νομίζω ότι όλες οι χώρες μέλη, από τη στιγμή που έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν συνυπογράψει την Ευρωπαϊκή Δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλοι όσοι μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είπαν τότε ότι θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από τον πόλεμο. Και πρέπει να το κάνουν λοιπόν, οφείλουν να το πράξουν σήμερα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γραμματικάκης τώρα από την Ελλάδα παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω ότι εσείς προσωπικά έχετε δείξει στο παρελθόν μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, παρόλο που καμιά φορά αυτό θεωρήθηκε ανάμειξη στα εσωτερικά μας και τώρα τα σημερινά νέα τα ξέρετε. Η Ελλάδα αγωνίζεται και σήμερα πληροφορούμε ότι είναι συνεπής της υποχρεώσεις της ως το προσφυγικό θέμα. Άλλοι σύμμαχοι Ευρωπαίοι υψώνουν τύχη, ενώ η Ελλάδα και πάλι, το ξέρετε, με τη συμφωνία του καλοκαιριού στην οποία είχατε ενεργό ενδιαφέρον, ε, πιέζεται ασφικτικά στην οικονομία της και ο ελληνικός λαός είναι θα έλεγα εξεγερμένος απέναντι σε αυτές τις διπλές ή τριπλές απειλές. Τι σκοπεύετε εσείς κύριε Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο ξέρω τις θέσεις του, να συστήσετε ή να αναμειχθείτε ή να επέμβετε για να ολοκληρώσετε το ενδιαφέρον σας για την Ελλάδα. From From Cyprus. Κύπρος τώρα. Η κυρία Κροκοκούμα. Και η δική μου ερώτηση αναφερόταν ε, στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε και βασικά ήθελα το σχόλιο μου α, ε, γινόταν σε σχέση με τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών της Ευρωζώνης που στην ουσία να κυνηγούμε να μεταλλαχτούν για να εξυπηρετούν δίθεν την ελεύθερη αγορά. Ε, και στην ουσία και την ηγεμονία της αγοράς, εντείνοντας έτσι τις κοινωνικές και εργασιακές ανισότητες. Αναφέρεται στην επισκόπηση ότι υπάρχει κάποια μείωση στην ανεργία, ε, χωρίς να γίνεται καμιά αναφορά και συσχετισμό σε σχέση με τη μερική απασχόληση που είναι πλέον η πλειοψηφία των εργαζομένων, χωρίς κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλες ε, μέτρα στήριξης. Για μας στην Κύπρο η κινητικότητα των εργαζομένων σημαίνει μετανάστευση. Είμαστε νησί και κινητικότητα σημαίνει μετανάστευση. Το λοιπόν, πώς μπορούν τα κράτη-μέλη να επαναχτίσουν το δικαίωμα χάραξης της δικής τους δημοσιονομικής πολιτικής που να έχουν και τον έντονο κοινωνικό χαρακτήρα που απαιτείται. Θα μείνω εδώ, αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα του κύριου Σούλτς ήταν διαφορετικό. From Portugal, Mr. Πορτογαλία, Τίκο Περέιρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Σούλτς. Δύο ερωτήσεις έχω. Όσον αφορά σημαντικά πράγματα για το μέλλον της Τραπεζικής Ένωσης και της Δημοσιονομικής Ένωσης. Ο μηχανισμός εγγύησης καταθέσεων είναι ζωτική σημασία για το μέλλον του ευρώ. Δεν προχωράει αρκετά γρήγορα όμω. οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι πιστεύει από αυτού. Δεύτερη ερώτηση, όσον αφορά τη Δημοσιονομική Ένωση και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση πολύ σημαντικά και αυτά για να αποφύγουμε την επόμενη κρίση. Όμως η επόμενη κρίση θα έρθει, δεν ξέρουμε, σε ένα, σε δύο, σε τρία χρόνια. Και δεν ξέρω κατά πόσο η Ευρώπη είναι προετοιμασμένη για την επόμενη κρίση ή θα οδηγηθεί στην καταστροφή τότε. Κωσυφοπέδιο, Πεκάη. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα. Γνωρίζω ότι όλοι στην Ευρώπη αγωνίζονται με τα οικονομικά προβλήματα και την οικονομική κρίση. Εγώ είμαι από το Κωσυφοπαίδιο. Κάποια οικονομικά προβλήματα και θέματα προοπτικής όσον αφορά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχουμε και εμείς. Στην ε, δικιά μας δημοκρατία επίσης πρέπει να προετοιμαστούμε καλύτερα και να προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε. Όμως η ελευθερία είναι κάτι πολύ βασικό για το κοσυφοπαίδιο και η ελευθερία είναι κάτι βασικό στις ρίζες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν έχουμε καλύψει τις προϋποθέσεις και προσβλέπουμε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ξέρω ότι μάλλον για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το σχολείο μου αυτό, αλλά αφού έφυγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λέω στον κύριο Σούλτ, γιατί ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας έχει στηρίξει πολύ. Ευχαριστώ. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τώρα ο κύριος Παπαδημούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι δεν είναι η ώρα για exit, όπως είπατε και στον κύριο Κάμερον. Είναι η ώρα για αποτελεσματικότερη και περισσότερη ευρωπαϊκή συνεργασία αλλά για, να είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία αποτελεσματική πρέπει όσα αποφασίζονται να εφαρμόζονται. Από το Σεπτέμβριο έχει αποφασιστεί και στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο η μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων αναλογικά. Μέχρι τώρα έχουν μεταγκατασταθεί περίπου 400. Πώς το σχολιάζετε και τι σκοπεύετε να κάνετε. Και επίσης, είναι δυνατόν η Ευρώπη να είναι ενωμένη αλλά να θέλουν οι Ούγγροι και οι Πολωνοί κονδύλια για τις αγροτικές επιδοτήσεις, χρήματα από τα διαφθορτικά ταμεία για τα έργα και σωστά και να αρνούνται την υπογραφή τους σε κοινέ αποφάσεις και στη συνθήκη του ΟΗΕ και στην ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αποφάσεις των Συμβουλίων. Πώς τα σχολιάζετε αυτά. From Poland, Πολωνία, κυρία Κλοκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε ερωτήσεις για την οικονομία. Οι πολιτικοί πρέπει να φροντίζουν να προχωράνε προς μια βελτίωση της οικονομικής κατάστασης. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο λοιπόν Στρατηγικών Επενδύσεων θα πρέπει να συνδυάσει τις δυνάμεις του με άλλα ταμεία. Πρέπει λοιπόν στην αναθεώρηση να απλοποιήσουμε τους κανονισμούς με τέτοιο τρόπο ώστε η συνέργεια να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και άρα να αποδώσουν περισσότερο όλες οι επενδύσεις, ιδιωτικές δημόσιε κλπ. Στο όνομα λοιπόν της Πολωνίας αλλά και ολόκληρης τη Ευρώπη μπορώ να πω ότι στην Πολωνία έχουμε προχωρήσει όσον αφορά την ανάπτυξη και η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που να βασίζεται σε πέντε πυλώνες, σε και καινοτομία, κεφάλαια για την ανάπτυξη, επέκταση και βιώσιμη ανάπτυξη. Επίση, θα πρέπει να προσθέσουμε εδώ και την ανάπτυξη τη υπαίθρου. Και έρχομαι στην ερώτησή μου. Ποια είναι η προοπτική για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να υπάρξει επαναβιομηχανοποίηση στην Ευρώπη. Τονίζονται μέχρι τώρα οι υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωτάω, είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και στη βιομηχανία, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που χρειάζεται η Ευρώπη σήμερα. Εν κατακλείδη, μία ερώτηση προς τον πρόεδρό μας. Ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκή Επίτροπή όσον αφορά το Nord Stream 2, τον αγωγό φυσικού αερίου. Ξέρουμε ότι παραβιάζει τον ελεύθερο ανταγωνισμό το σχέδιο αυτό και δεν ευθυγραμμίζεται με την αρχή της αλληλεγγύης. Τέλος. Θέλω να ρωτήσω και το εξής για τον άνθρακα. Μπορούμε να επεξεργαστούμε τον άνθρακα με διαφορετικό τρόπο έτσι ώστε να σωθούν χιλιάδες θέσεις απασχόλησης στην περιοχή από όπου προέρχομαι. Yes, thank you, Mr. President. And thank... Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για τα τόσο ξεκάθαρα λόγια σας που μεταξύ άλλων αναφερθήκατε στην ε, Συρία και είπατε ότι ο πόλεμος είναι εκείνος που οδηγεί τόσους ανθρώπους στην προσφυγιά. Με κάθε σεβασμό, την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίνατε ψήφισμα που λέει ότι τόσα έχει κάνει η ΝΤΑΣ είναι γενοκτονία. Αυτό όμως τι σημαίνει, ότι οι χώρες μας έχουν τώρα ανθρώπους οι οποίοι έχουν ε, φύγει από τις χώρες τους για να αποφύγουν αυτή τη γενοκτονία και εμείς δεν θέλουμε να τους αφήσουμε στις χώρες μας. Έπειτα η συνεργασία με την Τουρκία πώς προχωράει. Η χώρα τώρα ε, δέχεται κόσμο από τη Συρία και εμείς πληρώνουμε δισεκατομμύρια σε μια χώρα η οποία τελικά ε, δυναμητίζει τον πόλεμο στη Συρία. Εσείς πώς θα διασφαλίσετε ότι θα υπάρξει περισσότερη ειρήνη και ότι τελικά δεν πληρώνουμε για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην περιοχή αυτή του κόσμου. Καριέρα Ιταλία. Κύριε Καριόλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ε, κατάλαβα ότι μου δώσατε το λόγο, συγγνώμη. Πρέπει να καταλάβουμε αυτά ακριβώ που μας είπε ο πρόεδρος Σούλτς πριν από λίγο. Γιατί έδωσε την προτεραιότητα στην συνάντηση αυτή με τον ε, Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, τον κύριο Κάμερον ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ε, συζητήσει το θέμα ε, και του δημοψηφίσματος ε, ή και της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό είναι ενδεικτικό μιας ευρωπαϊκής κατάστασης που είναι σαφής. Εισακούεται μια χώρα μόνο όταν θέτει όρους και ιδίω όταν η χώρα αυτή είναι εκτός από την Ευρωζώνη. Εμείς είμαστε μια φωνή που πλέον είναι μοναδική στην Ευρώπη. Αρκετές ε, χώρες ε, ε, μιλούν προς την ίδια κατεύθυνση. Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή της συζήτησης στο θέμα του ευρώ. Οι σχέσεις των διαφόρων χωρών ε, αλλά και του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συζήτηση αυτή κάθε φορά προσπαθούν να αυξήσουν την διαπραγματευτική ε, σχέση όταν υπάρχει μια απειλή εξόδου είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από το ευρώ. Θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη σημασία σε αυτά τα φαινόμενα, τα οποία πλέον ε, είναι φαινόμενα τα οποία εμφανίζονται σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να ξεκινήσει και μια διαδικασία Εντό του Κοινοβουλίου για να γίνει μια σαφή συζήτηση για αυτή τη διάθεση αρκετών χωρών να αμφισβητήσουν ε, το ευρωπαϊκό όραμα. Ευχαριστώ. Από το Ηνωμένο Βασίλειο και πάλι η Βαρονή Φάλκνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μας δίνετε ε, και στοιχεία από τη συζήτηση σας με τον Πρωθυπουργό Κάμερον. Θα ήθελα να συνεχίσω από κάποια από τα σχόλια που κάνατε ε, την ανησυχία ε, των χωρών εντός και εκτός της Ευρωζώνης και με άλλα λόγια δηλαδή του Ηνωμένου Βασιλείου. Εμείς ως Ηνωμένο Βασίλειο θέλουμε να είναι επιτυχημένη η Ευρωζώνη. Θέλουμε η Ευρωζώνη να βγει από την ύφεση και να έχει οικονομίες οι οποίες ε, ε, έχουν καλά αποτελέσματα και να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για την ολοκλήρωση. Εγώ είμαι ε, υπεύθυνη πρόεδρος στην Επιτροπή στην έρευνα που κάνουμε. Ποτέ δεν μας είπε κανείς ότι θέλει να αποτύχει η Ευρωζώνη. Είναι προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι είστε εμπορικός μας εταίρος, γείτονας και το καθεξής. Ε, ήλπιζα λοιπόν επί τη ευκαιρία να πω και σε εσά κύριε Πρόεδρε και στους υπόλοιπους ευρωβουλευτές ότι ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις χώρες της Ευρωζώνης και παρακολουθούμε και την πρόοδό τους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δυστυχώς ο πρόεδρος Γιούνκερ δεν απάντησε στι ερωτήσει μου που σχετίζονταν με το θέμα αυτό, αλλά ήθελα να το διευκρινίσω αυτό από την ε, οπτική του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ. Τελευταίος ο πριν δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Γιάκομψον από τη Σουηδία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να τονίσω ε, ότι το θέμα το οποίο έφυξε η Αυστρία είναι αντίστοιχο με την κατάσταση στη Σουηδία. Οι Σουηδοί πολίτες και το Σουηδικό Κοινοβούλιο πραγματικά διαρωτώνται εάν ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έπρεπε να κάνει κατανομή ε, των προσφύγων στην Ευρώπη με τρόπο που να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς την κατάσταση των προσφύγων. Γιατί δεν έχει γίνει τίποτα από τότε που έλαβε τη σχετική απόφαση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν είναι καλό προηγούμενο όταν έχουμε τόσα πολλά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση επίσης. Ε, να μην αντιμετωπίζουμε προβλήματα από κοινού. Και ήθελα να πω σε όλους τους παρισταμένους ότι οι Σουηδοί δεδομένου ότι είναι και από αυτούς που συνεισφέρουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τώρα πλέον χρειάζονται ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και διαπιστώνουν ότι δεν λειτουργεί αποτελεσματικό. Δεν είναι εύκολα να μιλάς για μεγαλύτερη συνεργασία και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε μια χώρα σαν τη Σουηδία αυτή τη στιγμή. Έχουμε νέα προσωρινή νομοθεσία ασύλου, η οποία πλέον μας θέτει στο χαμηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης ε, προς την ε, ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό γίνεται γιατί το Δουβλίνο δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και τα άλλα κράτη-μέλη δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Κύριε Σούλτς, λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση. Έχει αποφασιστεί με την κατάσταση γιατί δεν λειτουργεί. Ευχαριστώ και τώρα για τα συμπεράσματα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Μάρτιν Σούλτ. Ευχαριστώ. Οι ερωτήσει σα αφορούν πολλά και διαφορετικά σημεία πολιτικής. που συνδέονται μεταξύ τους και αν δούμε και τις λεπτομέρειες των προβλημάτων και των άλλων των προβλημάτων έχουμε μια γενική εικόνα της δραματικής κατάστασης ε, στην οποία βρισκόμαστε ειδικά αυτή την εβδομάδα. Θέλω να είμαι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαλυθεί. Και εδώ στο Κοινοβούλιο υπάρχουν πάρα πολλοί που θα Χαιρόταν με μια τέτοια εξέλιξη. Όποτε είναι κάποιοι ότι όποτε είναι κάποιοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άχρηστη και κατά της λαϊκής βούλης κτλ. Από τα δεξιά σηκώνονται κάποιοι και χειροκορτάνε Και τα κόμματα αυτά στην Ευρώπη που λένε πως ε, το συμφέρον των εθνών ε, κατησχεί του συμφέροντος ε, της κοινότητας και ότι η δικιά μου χώρα είναι πιο σημαντική από άλλη, ότι η Ευρώπη είναι άχρηστη και πρέπει να αναδιαταχθεί. κερδίζουν τις εκλογές. Και έχουν μεγάλη στήριξη. Και επειδή με ρωτήσετε για την προσωπική μου άποψη, και είμαστε υπέρ της ε, εμβάθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε σοβαρή έντονη αντιπολίτευση. Ε, κάποιος βρίσκεται εδώ πέρα ε, Α, μόλις μπαίνει στην αίθουσα έδινε μόλις συνέντευξη στα ΜΜΕ και λέει πως έχει ήδη αποτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών είναι υπέρ της εμβάθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος είναι ε, ο οποίος μόλις ήρθε να δώσει μια συνέντευξη και έφυγε αμέσω. Εγώ είμαι υπέρ του να παραμείνουμε ενωμένοι. Να παραμείνει ενωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η ιστορική πείρα, ειδικά στην Ευρώπη, μας ε, διδάσκει ένα μάθημα. Όταν οι χώρες ε, και τα έθνη στην Ήπειρό μας δεν ε, συνεργάστηκαν διασυνοριακά, η Ευρώπη απέτυχε. Και το αποτέλεσμα ήταν καταστροφή για τα έθνη της Ευρώπης. Γι' αυτό το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, κατά την άποψή μου, ήταν η καλύτερη περίοδος στην ευρωπαϊκή ιστορία και βασίστηκε σε μία αρχή, στην αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών και εθνών. Και βασίστηκε στην αρχή ότι είμαστε πιο ισχυροί ενωμένοι. Και στο ότι βεβαίως υπάρχει η αμοιβαία αναγνώριση των διαφορετικών συμφερόντων. Αλλά το ότι είμαστε διατεθειμένοι να βρούμε μία δίκαιη συμφωνία είναι κάτι το επιτακτικό για να υπάρχει αξιοπρέπεια και ειρήνη και δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Οπότε για να απαντήσω σε όσους μίλησαν για τους πρόσφυγες. Η αλληλεγγύη είναι μια αρχή θεμελιώδης. Και όποιος λέει ότι εγώ είμαι αλληλεγγύος μόνο όταν με συμφέρει η αλληλεγγύη μου έχει προϋποθέσεις δηλαδή το δικό μου το συμφέρον, όποιος δεν βλέπει την αλληλεγγύη ως κάτι το αμφίδρομο, ότι κάτι παίρνεις και κάτι δίνεις. τότε πραγματικά ρίχνει, ε, εμποδίζεται τα γρανάζια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία, η Αυστρία, η Ελλάδα, η Σουηδία δεν μπορούν μόνες τους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Και έχετε δίκιο από τους 160.000, ε, ε, το είπε ο κύριος Παπαδημούλης, έχουν ε, μετακινηθεί 400 άτομα. Αλλά όταν λέει η Γαλλία 30.000 άτομα, η Γερμανία 40.000, έχουν 70.000 ήδη πάρει και απομένουν για τις υπόλοιπες χώρες 90.000 άνθρωποι. 2-3.000 σε κάθε χώρα δηλαδή. γίνεται αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το αδύνατο. Είπαμε να ληφθεί υπόψη το ΑΕΠ, ο πληθυσμός, το αριθμός των ανέργων σε κάθε χώρα και το πόσους έχει ήδη δεχτεί. Νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ δίκαιη ε, κλίδα κατανομής και πρέπει να δούμε ακριβώς την επιπτώση του προβλήματος, όχι να πηγαίνουμε σε ιδεολογικέ αντιπαραθώσει Και πρέπει να το λύσουμε αν δεν θέλουμε να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ερώτημα του, Ιτα... του Ολλανδού συναδελφού. Ναι, θα έχουμε και άλλε τέτοιε ε, ροέ προσφύγων. Και ξέρω πώ είναι δύσκολο να διαπραγματευόμαστε μια χώρα όπω ε, η Τουρκία, η οποία με την πολιτική τη ε, στους Κούρδους, και ξέρω πως είναι επίμαχο το θέμα εδώ μέσα, κάνει αυτά που κάνει, αλλά απ' την άλλη ως κάποιος ο οποίος έχω πάει συχνά εκεί πέρα, ξέρω πως οι πρόσφυγες οι Σύριοι στα τουρκικά στρατέποδα ε, είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι σε κάποια κρατημέλη της Ένωσης. Και είναι, θα έλεγα, υποδειγματική η κατάσταση εκεί πέρα. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω πως η Τουρκία είχε ανοιχτά τα σύνορά της με τη Συρία για μεγάλο διάστημα για να μπαίνουν πρόσφυγες. Και μπορείτε τώρα να, να δείτε. Ε, πράγματι, τους απευθύνω έκκληση όντω να ανοίξουν τα σύνορα στο Κίλης, ε, κοντά στο Χαλέπι, για να μπουν οι πρόσφυγες. Είναι πράγματι δύσκολο, γιατί χρειαζόμαστε την ε, Τουρκία για να ρυθμιστεί το, το ζήτημα. Υπάρχει λοιπόν η ηθική πτυχή την οποία αναφέρατε, εγώ θα σα απαντήσω ρεαλιστικά. Χωρίς συνεργασία της Τουρκία δεν θα μπορέσουμε να το λύσουμε το θέμα. Αυτό βεβαίω δεν σημαίνει ότι πρέπει να σιωπήσουμε. Πρέπει να ασκήσουμε και κριτική και να συνεργαστούμε. Και θεωρώ λοιπόν πως το ερώτημα του Σουηδού συναδέλφου απαντήθηκε. Τώρα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια και γρήγορα. Και ελπίζω να δεχτεί αυτή την ε, βοήθεια έχει μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κρίση και αντιμετωπίζει μια δραματική κατάσταση με τους πρόσφυγες. Αυτό δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει καμία χώρα μόνη της. Γι' αυτό πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα και στα hotspots και όσον αφορά την μετεγκατάσταση γιατί δεν έχει νόημα να φτιάξουμε ένα hotspot να, να έρχονται άνθρωποι και μετά να μην μπορούμε να τους ε, κατανείμουμε. Η Ελλάδα δηλαδή έτσι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα μεταβληθεί σε ένα τεράστιο στρατόπεδο υποδοχής προσφύγων. Ε, δεν το θέλουμε αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται κατεπηγόντως το σύστημα αυτό και ο Γάλλος Πρωθυπουργό είπε το Σάββατο πως η χώρα του ανεξαρτήτως ε, των υπολείπων ζητημάτων είναι διατεθειμένη να δεχτεί 30.000 πρόσφυγες Οπότε για να κατανείμουμε αυτούς τους 160.000 που είπαμε τώρα. Η αξιοπιστία βεβαίω τη Ευρωπαϊκή Ένωση χάνεται κάθε μέρα αν δεν είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε ε, αυτή την κατανομή που αποφάσισαν τα κράτη-μέλη όλα για την ε, Τραπεζική Ένωση και την εγγύηση των ε, καταθέσεων. Υπάρχουν εδώ πέρα όλοι οι ειδικοί ευρωβουλευτές. Να πω κάτι εγώ προσωπικά βρίσκονται και στην άλλη εδώ πέρα από την Γερμανία που είναι πάρα πολύ ακαθόδες στο θέμα και έχω και εγώ πράγματι και στενή σχέση με το σύστημα το γερμανικό των ε, ταμιευτηρίων ε, θα πρέπει όμως να βρεθεί μια ρύθμιση για αυτό το ζήτημα αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει στο να μην υπάρχει μια εγγύηση καταθέσεων στην Ευρώπη. Γιατί ο συνάδελφος από την Πορτογαλία, η συνάδελφος από την Πορτογαλία το είπε. Όταν έρθει η επόμενη κρίση και οδηγήσει πάλι στο να μην είναι σταθερές οι τράπεζες και να πρέπει πάλι να πληρώσει ο φορολογούμενος, δεν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και πολιτικά πλέον την κρίση. Μια τελευταία παρατήρηση για τη σύμβαση, για αυτά που είπατε για την γενοκτονία. Δεν θέλω... Θα με συγχωρήσετε τώρα, δεν είναι ότι δεν θέλω να απαντήσω, πρέπει να πάω στην διάσκεψη των πρόεδρων των ε, κοινοβουλευτικών ομάδων. Αλλά κοιτάξτε, τα κράτη θα πρέπει, τα κυρίαρχα κράτη θα πρέπει να δουν ε, ε, το τι θα κάνουν, γιατί ε, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρασε ένα ψήφισμα, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να το εφαρμόσει. Τώρα, η συνάλφος από την ε, Σιλεσία. Ναι, η απάντηση είναι σαφώς ναι. Χρειαζόμαστε την Ευρώπη βιομηχανοποιημένη. Αλλά το μέλλον της ε, βιομηχανίας και των υπηρεσιών ε, που συνδέονται με την βιομηχανία εξαρτάται από την ψηφιακή μας αποτελεσματικότητα. Λοιπόν, η ψηφιακή εξέλιξη είναι η άλλη πτυχή του νομίσματος. Ε, όσον αφορά τώρα τον άνθρακα, εγώ προέρχομαι από μια τέτοια περιοχή η οποία είδε το κλείσιμο των ανθρακοριχείων και πέρασε ένα μετασχηματισμό που κράτησε 30-40 χρόνια. Οπωσδήποτε κάποιες ε, περιοχές θα υποφέρουν για να πάει η Ευρώπη σε ένα μέλλον χωρίς άνθρακα. Γι' αυτό αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να αποφύγουμε να υπάρξει ολόκληρη κατάρρευση οικονομικών κλάδων και περιφερειών. Το έχουμε καταφέρει σε άλλες περιφέρειες, αλλά πρέπει να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και κάνει και στο παρελθόν. Θα πω ένα πράγμα, ποιος ξέρει μια τέτοια περιοχή, ξέρει πως δεν γίνεται η αλλαγή αυτή από τη μια μέρα στην άλλη, μια διαδικασία μακροχρόνια. Λοιπόν, ε, μπορεί να μην απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Με συγχωρείτε, πρέπει να ξαναφύγω. Υπάρχουν όμως εδώ πέρα πολλοί συνάδελφοι που για τα θέματα του κοσφοπεδίου, της Τραπεζικής Ένωσης, του Νόρστροιν Stream και της ε, Ευρωζώνης νομίζω τα ξέρουν ε, εξίσου καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ Μάρτιν. Και τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο γύρο. Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο Μοσκοβισή, ο οποίος θα συμμετέχει σε αυτή τη δεύτερη συνεδρία της Ολομέλειας ως Ευρωπαίος Επίτροπος Αρμόδιος Οικονομισματικών και Νομισματικών Θεμάτων, Φορολογίας και Τελωνίων. Η συνεδρίαση θα έχει ως πρόεδρο τον κύριο Τόμας ε, Χάνταλ, πρόεδρο της Επιτροπής ε, ε, Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΟΝ θα αντικαταστήσει τον κύριο Γκουαλτιέρη, ο κύριος Μάρκος Βέμπερ θα είναι εδώ, λόγω ε, της έκτακτης συνεδρίασης της διάσκεψης των Προέδρων. Ο πρόεδρος δεν μπορεί να παραστεί, όπως σας είπε και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Οι πολιτικές ομάδες για την ε, ε, διαπραγμάτευση με το Ηνωμένο Βασίλειο εργάζονται πισταμένα και χρειάζονται φυσικά ε, τον κύριο Γκαλτέρη. Ευχαριστώ πολύ και καλή τύχη. <laughs>